αύριο. Θα ήθελα να σε ενημερώσω όλους ότι η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο 5η 19η Ιανουαρίου του 2017 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και μετά από τις 3 μέχρι τις 4. Το πρόγραμμα, η ατζέντα είναι στην